So, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls Sie noch einen Platz finden, setzen Sie sich bitte hin. Und wir können dann anfangen mit Μπορούμε να αρχίσουμε με την προετοιμασία της 19ης Συνόδου από, που θα αρχίσει στις 11 του μήνα στη Βαρσοβία, Πολωνία και Έχουμε μαζί μας ε, τον ε, μελλοντικό πρόεδρο της ΚΟΠ. Ε, θα κάνουμε μια μικρή προετοιμασία. Και βεβαίως σας έχουμε μεταδώσει και το άλλο μήνυμα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα, πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ πέρα την δουλειά μας. Έχουμε ένα ψήφισμα που προετοιμάζουμε. Ελπίζω να υπερψηφιστεί, αλλά βεβαίω εντάξει δεν έχουμε φτάσει εκεί πέρα ακόμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τα προφορικά ερωτήματα. Το ψήφισμα λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Αλλά πριν ε, δώσω τον λόγο συναδέλφους, στον συνάδελφο εν πάση περιπτώσει, στον συνάδελφο. Ε, Καλωσορίζω τον κύριο Ρέτσκα, Διευθυντή διεθνών σχέσεων και κλιματικής στρατηγικής στη Γενική Διεύθυνση Κλίματος. Και θα μας κάνει μια εισαγωγή και μετά ξεκινάμε. Έχετε λοιπόν το λόγο αγαπητέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και ε, να πω λίγα λόγια για τη Βαρσοβία. Θα συνεχίσω τώρα στα αγγλικά, μια γλώσσα την οποία ξέρω κάποιος καλύτερα. Η Βαρσοβία Στη Βαρσοβία μάλλον θα γίνει μια δύσκολη διάσκεψη, κυρίως ως προς ε, την κοινή γνώμη, διότι στη Βαρσοβία δεν περιμένουμε ε, κανένα νέο πρωτόκολλο του Κιώτο ή κάποια συμφωνία της Κοπενχάγης ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο συναρπαστικό, αλλά είναι ένα βήμα προς την επίτευξη της συμφωνίας που ελπίζουμε να συναυθεί στο Παρίσι το 2015. Παρ' αυτά θα είναι σημαντική σχετική διάσκεψη διότι θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε συμφωνία όπως έλεγα μετά από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο Παρίσι το 2015. Βλέπω, ε, εν ώψη λοιπόν αυτής της συμφωνίας συνειδητοποιούμε ότι όλα τα συμβαλόμενα μέρη έχουν αρχίσει να σκέφτονται ακριβώς ποια θα είναι η συμβολή τους σε αυτή τη συμφωνία το 2015. Ίσως θα έχετε ακούσει ότι υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος σε σχέση με το περιεχόμενο ακριβώς συμφωνίας του 2015. Ξεκάθαρα επικρατεί η άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχουν δεσμεύσεις, νέες δεσμεύσεις ε, που υπερβαίνουν την περίοδο μέχρι το 2020. Αλλά ε, αυτό δεν προδικάζει την έκβαση των διαπραγματεύσεων γιατί κάποια συμβαλόμενα μέρη πιστεύουν ότι θα έπρεπε ενδεχομένω μεταγενέστερο στάδιο να το επιδιώξουμε για την ακόμη πρόωρο. Πάντω είναι ένα ε, εφαλτήριο, δηλαδή ένα σημείο προβληματισμού για τα συμβαλόμενα μέρη σε σχέση με τη μελλοντική του συμβολή για το 2015. Ξέρετε ότι ο πρόεδρο Βαρόσο και η Επίτροπος Χέντεγκαρτ έχουν αναλάβει δέσμευση να εξετάσουν ε, την ε, μελλοντική κατάσταση της περιβαλλοντικής πολιτικής μέχρι το 2030. Ε, και αυτή είναι και η απαρχή μιας ευρωπαϊκής εντολής για τη σύναψη της συμφωνίας του 2015. Περί τα τέλη του τρέχοντος θα έχουμε μάλλον το σχέδιο της θέσης του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να συζητηθεί και εδώ στο Κοινοβουλίο και στα κράτη-μέλη με απότερο στόχο να διαμορφωθεί, να παγιωθεί η θέση της ΕΕ για τη Συμφωνία του 2015. Ε, και ξεκαθα... Ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ε, στη διάσκεψη της Βαρσοβίας προς όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Επίσης, ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να διαπιστώσουμε ποιοι χρειάζονται τεχνική αρρωγή για να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να αποφασίσουν κατά πρώτον ποια θα είναι η συμβολή τους στη η συμφωνία του 2015. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεύτερο. κάτι που είπαμε και σήμερα το πρωί, όταν ακούσαμε τους υπουργούς, υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα που μας χωρίζει από το 2030, από το 20 μέχρι το 30. Βάσει τη εντολή του Durban, ε, όλα τα συμβαλόμενα μέρη πρέπει να εξασφαλίσουν τη γεφύρωση αυτού του χάσματος προσδοκιών και οι ε, λιγότερα αναπτυγμένες χώρες και οι μικρές νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες απευθύνουν έκκληση το 2014 να αναδειχθεί σε έτος φιλοδοξίας, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να αναλογιστούν ποιοι είναι οι δικοί τους στόχοι που έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν μέχρι το 2020. Δύσκολη συζήτηση λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλεφθεί στη διαδικασία να ε, επί τη βάση του πρωτοκόλλου του Κιώτο για τα συμβαλόμενα μέρη. Αλλά για τα μέρη που δεν είναι συμβαλόμενα στο πρωτόκολλο του Κιώτο δεν προβλέπεται τίποτα. Και ξέρετε ότι το 30% είναι υποαίρεση. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και ποιες είναι αυτές μεταξύ άλλων ότι όλα τα συμβαλόμενα μέρη πρέπει να ε, αναλάβουν δέσμευση, να κάνουν κάποιο pledge. Οπότε Χρειαζόμαστε ένα εξισερωπημένο αποτέλεσμα στη Βαρσοβία, ούτως ώστε το 2014 να μην, βρεθεί, να μην δεχθεί επιθέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Ε, ας περάσω σε ένα άλλο τομέα, τον τομέα της εφαρμογής. Η δημόσια γνώμη μάλλον έχει ξεχάσει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν ληφθεί πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ε, ανέκαθεν έλεγα πως Πλέον έχουμε κλείσει ένα κεφάλαιο στις διεθνείς περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις. Αυτά που θέλαμε στην Κοπενχάγη τα πετύχαμε τα περάσμενα χρόνια. Χρειαζόμαστε ισχυρότερες δεσμεύσεις από περίπου 19 χώρες ε, του κόσμου που καλύπτουν το 80% των παγκοσμίων εκπομπών. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εισερχόμεθα σε μια νέα φάση δεσμεύσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιώτο και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει όλα τα έγγραφα για να κυρωθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό απαιτεί ε, κύρωση από πλευρά των 28 κρατών μελών στα εθνικά τους κοινοβούλια. Ε, η διαδικασία αυτή λοιπόν έχει ως εξή, θα μας ρωτάνε οι υπόλοιπε χώρε του κόσμου μέχρι που έχουμε φτάσει. Λοιπόν η απάντηση είναι ότι από τις αρχές του 2013 έχουμε αρχίσει την εφαρμογή και θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει δυνάμει του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤ. Πέραν αυτό. Θέλουμε αντίστοιχε προσπάθειες και σοβαρότητα ω προς την εφαρμογή να δείξουν και τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη ε, και στη Βαρσοβία συγκεκριμένα. Δηλαδή όσα τα συμπεφωνημένα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υλοποιούνται. Και αυτό ισχύει και για κάποιους ε, νέους οργανισμούς, το Ταμείο για το Πράσινο ε, Κλίμα, το, το, το, Ταμείο για τη Χρηματοδότηση, το Κέντρο για τις Καθαρές Τεχνολογίες, το αντίστοιχο δίκτυο και το καθεξής. Όλα αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν στη Βαρσοβία και να αποφασίσουμε τα οργανογράμματα και τα προγράμματα εργασίας αυτών των οργανισμών Μόνο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και εμεί να έχουμε αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μα για να αποφασίσουμε τη συμβολή μα. Ένα από τα δυσχερέστερα ερωτήματα που θα μα απασχολήσουν είναι η χρηματοδότηση. Έχουμε τι δεσμεύσει τη Κοπενχάγη για κινητοποίηση 100 δις αμερικανικών δολαρίων από πλευράς του ανεπτυγμένου χώρου, ε, ε, κόσμου συγγνώμη, μέχρι το 2020 για τη χρηματοδότηση αυτής της πολιτικής. Κάποιες χώρες μας ζήτησαν να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι προθέσεις μας, τα σχέδιά μας για την κλιμάκωση των προσπαθειών, ώστε μέχρι το 2020 να επιτύχουμε ε, το στόχο του συνολικού όμως πόσου. ξέρετε στις δημοσιονομικές διαδικασίες και εδώ στο Κοινοβουλίο ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει η συγκεκριμένη πρόταση μέχρι να φτάσουμε στο 2020. Δεν είναι εύκολο ούτε για την Επιτροπή ούτε για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Αυτό που σίγουρα πρέπει να δείξουμε από πλευρά Ένωση είναι ότι αποκρινόμαστε στα αιτήματα των ε, αναπτυσσομένων χωρών, ώστε και εκείνε να μπορέσουν να τηρήσουν τι δεσμεύσει συμφωνία τη Κοπενχάγη και τα όσα ακολούθησαν. Τα κράτη-μέλη κοιτάζουν τα λογιστικά του βιβλία επισταμένα για να μπορέσουν να πούν υπάρχουν ε, κάποια πράγματα σε σχέση με το τι κάνουμε το 2013 για τη χρηματοδότηση και τι σκοπεύουμε να κάνουμε ε, μέχρι το 2020. Μία συγκεκριμένη συνιστόσα είναι το Ταμείο Προσαρμογής. Θα δείτε ότι θα αποκτήσει ιδιαίτερο ειδικό βάρος σταδιακά, διότι αυτό είναι συνάρτηση της μόχλευσης του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης. Όσοι γνωρίζετε τι γίνεται ε, στην αγορά του διοξιδίου του άνθρακα θα γνωρίζουν ότι υπάρχει πολύ χαμηλή ζήτηση για αυτούς τους πόντους, στα credits, ε, οπότε δεν θα έχουμε εισοδήματα για να ε, χρησιμοποιήσουμε τη μόχλευση του μηχανισμού καθαρή ανάπτυξη και κυρίω αναπτυσσόμενε χώρε παραπονιούνται ότι στο Ταμείο Προσαρμογή δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια. Κάποια κράτη-μέλη θα θέλουν σε θελούσια βάση να αναλάβουν δέσμευση για το Ταμείο Προσαρμογή. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα υπάρχει δέσμευση να συνεχίσουμε την ε, ε, κλιμάκωση τη χρηματοδότηση για το Ταμείο Προσαρμογή, αλλά προ το παρόν όλα αυτά εντάσσονται στο συνολικό τροπλαίσιο των συζητήσεων του επομένου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι βαριά η μερίσια διάταξη τη ΚΟΠ στη Βαρσοβία, πολλά τεχνικά ζητήματα αλλά και κάποιε πολιτικέ μάχε. Ο μεγαλύτερο φόβο από πλευρά μα είναι ότι η συζήτηση περί χρηματοδότηση θα μπορούσε, θα μπορούσε κάποιος να τη χρησιμοποιήσει ούτω ώστε ε, να κρατήσει κάποιες χώρες ο μύρος εν ώψη της συμφωνίας ε, του 2015 διότι ε, είναι σίγουρο ότι κάποια πράγματα δεν θα μπορέσουμε να τα διεκπαιρεώσουμε μέχρι τότε και θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε ε, συμμάχους από τους αναπτυσσόμενους χώρους, από την ομάδα της Αφρικής, από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για να υπάρξει συσπήρωση αλλά και αξιόπιστες απαντήσεις στις ερωτήσεις που μας κάνουν για τη χρηματοδότηση της πολιτικής μας τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε και τη γενική εικόνα που μας δώσατε. Οπωσδήποτε θα είμαστε παρόντες με μια αντιπροσωπεία στην Βαρσοβία και νομίζω πως πρέπει να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη να το χρηματοδοτήσουν το θέμα σοβαρά προσθέτουν διάφορα ποσά και αυτό κατέστη σαφές τυχαία όταν ε, είχαμε μια άλλη διεθνή αντιπροσωπεία. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λέμε στο κοινό. Οπωσδήποτε η άσκεψη θα είναι πάρα πολύ σημαντική και κάποια θέματα και το θέμα της χρηματοδότησης είναι σημαντικά. και για την πολιτική δράση, γιατί είναι καλά τα ψηφίσματα, αλλά ε, βεβαίω αν δεν κάνουμε τίποτα μετά δεν υπάρχει και αξιοπιστία. Δηλαδή υπάρχει αυτό το, το δικό μου το θέμα, το εμπόριο εκπομπών, αλλά υπάρχει και η καταπολέμηση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ξεκινάμε λοιπόν με τους ε, συνεισηγητές. να σας αυτούς και εγώ. Ο Καλ Χάιντς Φλόρεντς ήταν εκεί νομίζω. Από το 92. Καλ Χάιντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Χέμεν Μούντινγκ, ένα νεαρό ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα και βλέπετε πως έχει δώσει πάρα πολλές ε, μάχες για το θέμα. Είναι παλαιός ε, φίλος και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Δεν είναι βεβαίως βουλευτής του έλκα, αλλά του επέτρεψα κατ' εξαίρεση να έρθει. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Ναι, εδώ πέρα όμως αισθάνεται πιο άνετα. Τι να κάνω. Δεν φταίω εγώ. Ναι, δεν θα μείνει μόνιμα, μη φοβάστε. Κοιτάξτε, εμένα μου προξένει σε έκπληξη αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν για το τι ακριβώς συνεισφέρουμε. Αυτό είναι σημαντικό και για την εθνική μας πολιτική. γιατί βεβαίως το θέμα είναι αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν ξέρουμε πού πηγαίνει η Κομισιόν και πού θέλει να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα προσπαθήσουμε όπως πάντα να εργαστούμε επικοδομητικά, θετικά τα άλλα που αναφέρετε τώρα είναι διαφορετικά, αλλά κοιτάξτε, ο παγκόσμιος χάρτης έχει αλλάξει και χρειαζόμαστε ένα νέο κλιματικό πακέτο. Το αυτό το οποίο είχαμε μέχρι τώρα. Και το ερώτημα είναι, οι δομές μήπως που έχουμε εντός του ΟΗΕ, μήπως έχουν ξεπεραστεί. Πώς είναι δυνατόν με 195 χώρες να έχουμε ομόφωνα ψηφίσματα. Το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ είναι πολύ καλό παράδειγμα. Είναι ένα διαφορετικό σύστημα με καλά αποτελέσματα. Ε, και δεν είναι τόσο ευχάριστη η απλή κατάσταση. Ε, έτσι είναι η ζωή, δεν είναι ευχάριστη. Κοιτάξτε, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιες ομάδες ε, θα, θα έχουν πιο πλαίσιο. Μετά το πράσινο κλιματικό ταμείο, πάλι ο πρόεδρος λέει πως πρέπει να ρεύσουν ε, λεφτά και μάλιστα ρευστό. Τι νομική μορφή θα έχει μια τέτοια σύμβαση, μπορεί κάποιος να προσφύγει εναντίον της. Αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος. Θεωρώ λοιπόν πως οι ευέλικτοι μηχανισμοί, οι καθαροί μηχανισμοί ανάπτυξης ήταν κάτι που υποστήριζα στο παρελθόν, αλλά τώρα είχαμε αρνητικές εμπειρίες με τα MRV. Τι γίνεται, πώς τα μετράμε. Πρέπει λίγο να το δούμε. Ακούσαμε ήδη σήμερα για το ρόλο της ε, Προεδρίας ε, και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει κάποια όθηση από την Προεδρία. Το Μεξικό ήταν πολύ καλό παράδειγμα και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα η νέα έκθεση του IPCC να μας δώσει νέα στοιχεία. Και τέλος. καλό είναι να μην παθαίνουμε κατάθλιψη. Υπάρχουν χώρες και η υπηροί που είναι τόσο καλοί και εργατικοί όσο εμείς και με αυτές πρέπει να συνεργαστούμε. Νότια Κορέα, Αυστραλία. Ε, και έτσι θα αποκτήσουμε κάποιο βάρος. Χωρίς, χωρίς αυτό το δικό βάρος δεν θα γίνει τίποτα. Σας ευχαριστούμε. Νταν Γιώργενσεν δεν είναι εδώ. Ζητάει συγγνώμη. Μου έχει δώσει ένα σχόλιο. Γενικό σχόλιο λέγεται. Παρά το ότι οι προσδοκίες μας είναι περιορισμένες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να αυξήσουμε την πίεση για κλιματική δράση στο διεθνές πολιτικό σύστημα. Δεύτερον, να φροντίσουμε πως τα αποτελέσματα της ΔΟΧΑΣ ε, δεν θα εξασθενήσουν. Και τρίτον, και σημαντικότερο, να στηρίξουμε την πρόοδο προς μια παγκόσμια κλιματική συμφωνία 2015. Οπότε, δύο σημεία είναι σημαντικά. Η, η αύξηση της φιλοδοξίας, έτσι ώστε να φτάσουμε το 2020 σε μια δέσμευση εντός του ορίου των δύο βαθμών δεύτερων. Η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να δει το θέμα της αποδάσωσης και της έμεσης ε, χρήσης γης. Αυτά είναι τα σημεία που ήθελε να πει ο Νταν Γιόργενσεν. Και οπωσδήποτε ε, θα το δούμε στην διαπραγμάτευση. Κορίν Λεπάζ για την Άλντε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσα είπαν οι προηγούμενοι μιλητές, ε, συμφωνώ με αυτά. Εδώ αρκετοί συμμετείχαμε σε όλες τις συναντήσεις από την Κοπεχάγη από ο Καλχάινς και πριν μάλιστα. Και να σου το πω ειλικρινά, ειλικρινά. Κάθε φορά αισθανθήκαμε μια κάποια απογοήτευση. Και άλλωστε αυτό τονίζεται στο ψήφισμα η αντιπροσωπεία μας. Ε, είναι, την κρατάνε σε απόσταση μακριά από τις διαπραγματεύσεις. Και η εντύπωσή μας είναι η τελική κατάληξη είναι το ελάχιστο δυνατό για να οργανωθεί μια καινούρια. Και τώρα με άλλες αντιπροσωπείες να δούμε πού θα ενδεχόμενα θα είχαμε μια κοινή άποψη και να σχηματίσουμε μια ομάδα πίεσης υπέρ μια συγκεκριμένη εξέλιξη για το όλο θέμα. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Και να μην ζούμε μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Έχαμε τρεις κόπλου τη μία μετά την άλλη. Μιλάμε για το δισεκατομμύρια δολάρια, ναι, για το 2020 με καινοτόμες χρηματοδοτήσεις. Αυτές αναφερόμαστε, αλλά δεν λέμε ποιες είναι αυτές. Εντάξει, συζητάμε τώρα πόσοι εκπρόσωποι από τη μία ή την άλλη χώρα, σε τι επίπεδο κλπ. Υπέροχα όλα αυτά. Αλλά τι γίνεται, χωρίς χρήματα δεν εξυπηρετούν σε τίποτα αυτά. Και ιδιαίτερα συγκεκριμένους στόχους θα πρέπει να θέσουμε η Ευρώπη και το Κοινοβούλιο ενισχυμένοι θα έβγαιναν. Ίσως ε, πιο λιγότερο γενικές ιδέες παγκοσμίου χαρακτήρα, αλλά τουλάχιστον συγκεκριμένα με τους στόχους που θα πρέπει να πετύχουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε για την επισκόπηση κατάστασης για να ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι επαναστατικού χαρακτήρα η σύνοδος της Βαρσοβίας. Μπορεί κάποιοι να το επιθυμούν μεταξύ των οποίων και ο υπεφαινόμενος αλλά δεν θα είναι. Ελπίζουμε πάντως να ε, πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε σιγά σιγά τη συμφωνία του 2015 με τι εξελίξεις ε, στη Βαρσόβια και κάποιοι συνάδελφοι έχουν αρχίσει να κουράζονται με αυτέ τι συνόδου κορυφή για το κλίμα. Ε, οφείλω να πω ότι θα αυξάνονται διαρκώ οι προσδοκίες, θα μα παρακολουθεί ο κόσμο. εν ώψη τη συμφωνία του 2015 βέβαια. Αυτό είναι καλό γιατί μέχρι το 2009 είχαμε υψηλέ προσδόκίε και στη συνέχεια έχουμε ακολουθήσει ένα αρνητικό κύκλο θα έλεγα. Ε, και τώρα σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει η διάθεση και οι, εμείς οι ίδιοι και αυτό πρέπει να γίνει γιατί πρέπει να δείξουμε κάτι απτό μετά το 2015. Δεν μπορούμε απαθείς ε, να μην περιμένουμε τίποτα, να μην προσδοκούμε τίποτα, γιατί ε, το ίδιο θα συμβεί και για όλους τους υπόλοιπους αν το κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο επάξον την ευκαιρία που έχουμε και σίγουρα θα είναι από τις δυσκολότερες διασκέψεις, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε τη σύνοδο του Παρισιού, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να στεφτεί με επιτυχία. Και υπάρχουν και τα μεγάλα ερωτήματα. Τι μάθαμε από την Κοπενχάγη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό που ε, κανονικά θα έπρεπε να έχουμε μάθει είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τελευταία στιγμή μέχρι να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι φέτος στη Βαρσοβία θα πρέπει τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε σχέση με το πώς θα διαμορφωθεί η διαδικασία μέχρι το 2015. Δύο χρόνια υπολείπονται. Σε δύο χρόνια μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα, αλλά όχι αν απαθής περιμένει κανείς ε, ότι θα συμβούν ε, με μαγικό τρόπο τα πράγματα και το 2014, ε, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας Μπανκιμούν, πρέπει να είναι ένα... Ε, πλατή στο το οποίο θα ανέβουμε και θα αρχίσουμε ε, να ε, προσεγγίζουμε το 2015 για να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα καταθέσουμε και τις προτάσεις μας για τις δεσμεύσεις. Αν περιμένουμε το 2014 μέχρι να αρχίσουμε να ακούμε υποσχέσεις, τότε ξέρουμε ότι θα είναι μια νέα Κοπενχάγη το Παρίσι. Το 2014 οι προσφορές των συμβαλωμένων μερών πρέπει να είναι στο τραπέζι, ούτως ώστε να γίνει διαβούλευση με τους ε, εμπειρογνώμονες ε, για να δούμε ποιοι πρέπει να κάνουν ε, μεγαλύτερες προσπάθειες. Ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον αυτό. Αν αποτελματωθούμε σε μια συζήτηση για τη χρηματοδότηση και παγιδευτούμε σε αυτή, γιατί αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελοχεύει, δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Ένα άλλο στρατηγικό ζήτημα είναι όχι τι μάθαμε από την Κοπεχάγη, αλλά τι μάθαμε από την Τόχα μία από τις επιτυχίες της συνόδου ήταν αυτή της Ντόχα ακριβώς διότι έγινε ένα συνασπισμό με την Αφρικανική Ένωση και με τις ε, νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε η Κίνα, η Ινδία, η ΙΠΑ πίεση για να ε, προχωρήσουν. Και για αυτό δεν άκουσα απάντηση. Ξανακάνω την ερώτηση. Τι μπορεί η Ευρώπη να προσφέρει σε αυτά τα μέρη του κόσμου, κυρίως ε, στη στις νησιωτικές, ε, λιγότερο ανεπτυγμένες ε, χώρες ε, και την Αφρικανική Ένωση για να αποδείξουμε ότι είναι πιο φιλόδοξο το σχέδιο γιατί αλλιώς δεν θα μας πιστέψουν, θα πούνε ότι είναι μόνο λόγια και ευχολόγια αλλά στην πράξη δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πώς στη Βαρσοβία μπορούμε να κατοχυρώσουμε λοιπόν την αξιοπιστία μας ενώπιον αυτών που χρειαζόμαστε, τους χρειαζόμαστε, να πρέπει να συνασπιστούμε μαζί τους για να μπορέσουμε να πιέσουμε συνέχεια την Κίνα, την Αμερική και την Ινδία. Ε, και στο Ντέρμπαν ε, μας είχε απασχολήσει το ίδιο θέμα και στην Τόχα δεν είχαμε ακριβώ το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα δούμε λοιπόν πώ μπορούμε να το χειριστούμε στη Βαρσοβία. Ε, αυτή την τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντα, θα έλεγα ότι ο κινησμός που επικρατεί για τις κλιματικές αλλαγές, το σχολιάσατε, η IPCC την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιεύσει νέα έκθεση που συνθήκε. συνθήκες, οπότε όλες οι απόπειρες άρνησης, ε, όσοι παίζουν το χαρτί ότι δεν ε, υπάρχουν κλιματικές αλλαγές, ε, θα, δείτε, θα δουν στην έκθεση τις επόμενες εβδομάδες ότι ο στόχος των δύο βαθμών Κελσίου είναι το ελάχιστο στο οποίο πρέπει να αποσκοπούμε και ότι είναι υπαρκτές οι κλιματικές αλλαγές και αυτό θα θα μας οδηγεί σε μεγαλύτερη φιλοδοξία για όλα τα κράτη-μέλη μεμονωμένα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η επιστήμη θα μας προσφέρει τα τεκμήρια την επόμενη εβδομάδα εκ νέου και μόλις έχουμε αυτό στα χέρια μας πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι πιθανή μια θετική έκβαση το, στο Παρίσι το 2015. Πρέπει να το πιστέψουμε για να συμβεί. Αλλιώς ε, ο αρνητισμός ε, θα μας κάνει να πάρουμε την κατηφόρα και δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Πολύ σας ευχαριστούμε. Κρήτον Αρσένης και μετά Τζολάινεν. Ε, ευχαριστώ. Πολύ καλή ανάλυση του κύριου Ρούγκε Μέτσα. Στη Βαρσοβία πάλι θα μας επιτεθεί ο τύπος και θα μας παρακολουθεί στενά. στο Ντέρμπαν καταφέραμε να πείσουμε τους συμμάχους μας και δημιουργήσαμε αυτό το συνασπισμό που οδήγησε σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στο Ντέρμπαν ε, ε, σε πείσμα όλων των προβλέψεων. Αλλά και πάλι όμως δεν είχαμε ε, το αποτέλεσμα που θέλαμε και γι' αυτό στην Τόχα δεν είχαμε τόσο καλά αποτελέσματα όπως στο Ντέρμπαν. Τώρα και πάλι θα ασκηθεί πίεση σε εμά για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα... Εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ηγετικό ρόλο, νομοθετούμε, ε, πιέζουμε την ε, βιομηχανία μας. Και παρότι ε, ίσχυε και αυτό το 2009 στην Κομεχάγη, έχουν περάσει στο μεταξύ δύο χρόνια, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. 90 χώρες στον κόσμο, όπως βλέπουμε ετησίως εξάλλου, ε, στους, στις ε, συσκέψεις των παγκοσμίων νομοθετών, ε, σε όλες τις κόψεις δηλαδή, νέα νομοθεσία έχει εγκριθεί, φιλόδοξη νομοθεσία για την κλιματική δράση στα κοινοβούλια αυτών των 90 χωρών. Δεν είμαστε οι μόνοι δηλαδή που έχουμε να παρουσιάσουμε θετικά αποτελέσματα για την νομοθεσία και οι άλλοι έχουν πράγματα να δείξουν. Δεν είναι αρκετά καλή η φήμη μας, για να το πω. Απλά θέλουν, περιμένουν από εμά συγκεκριμένα πράγματα, η χρηματοδότηση, Δεσμεύσει. Θα είμαστε εκεί λοιπόν και θα μπορέσουμε για τα MRV, για τα LSF να τους δώσουμε ε, συγκεκριμένη πρόοδο για τα φθοριούχα αέρια, για όλα, πολλά πράγματα. αλλά θα περιμένουν ξαναλέω κάτι συγκεκριμένο. Γιατί υπάρχουν νομοθετικές εξελίξεις σε πάρα πολλέ χώρες. Εάν αποτύχουμε και δεν ανακτήσουμε την ε, εμπιστοσύνη των ε, συμμάχων μας, ε, την εμπιστοσύνη που κερδίσαμε ξαναλέω, εάν λοιπόν αποτύχουμε, τότε ενδέχεται να είναι αρνητικά τα αποτελέσματα της ε, Βαρσοβίας ε, ε, και αυτό αμαυρώνει και όλες τις προοπτικές για το Παρίσι το 2015. Είναι κέρια σημασία λοιπόν η Βαρσοβία και θα συμφωνήσω και πάλι με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Πρέπει ξεκάθαρα να κάνουμε βήματα προς αυτό το θεματολόγιο του 2015. Πώς, με ποιο τρόπο θα αρχίσουμε να δείχνουμε κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με τις δεσμεύσεις και τι θα γίνει καθοδόν μέχρι το 2015. Με ποιο τρόπο. Ήδη το 2014 θα είμαστε προετοιμασμένοι για ε, την πιθανή έκβαση του 2015 να φαίνεται ως το πιο πιθανό σενάριο. Αλλιώς θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε και για να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένα πράγματα χρειαζόμαστε ευφιέστερους τρόπους ε, λειτουργίας. Ε, Οπότε θα καταθέσω εγώ σχετικέ τροπολογίε στην Επιτροπή μα. Ευχαριστούμε, Κρήτονα. Ε, Τζολάινεν. Ε, ναι, ευχαριστώ. Κοιτώντα το περσινό ψήφισμα και το φετινό, θα μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη και να γράψουμε Βαρσοβία. Τα θέματα είναι ίδια. Το, το κλιματικό ταμείο είναι άδειο. το κενό των εξακολουθεί να υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διατηρήσει κάποια επιρροή στη διαδικασία. Φοβάμαι πως υπάρχουν δυνάμεις που δεν το βλέπουν επίγον το θέμα και καθυστερούν τη διαδικασία. Δεν ξέρω να ρωτήσουμε λοιπόν τον πρόσωπο της Κομισιόν αν ξέρει, αν νιώθει κάτι τέτοιο. Χώρες που λένε εντάξει τι βιαζόσαστε με το 2015, έχουμε μέχρι το 2020. Δεν ανάγκη να τα κάνουμε όλα στο Παρίσι, θα υπάρξει και επόμενη διάσκεψη. Πρέπει να τονίσουμε το κατεπήγον του πράγματος. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αντιθέτως, έχουμε χάσει ήδη πολύ χρόνο. Στο κενό των γιγατόνων το θέμα είναι τι προσφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίσαμε το 2020 το Κοινοβούλιο πάντα σε Κανκούν, Ντέρμπαν και Ντόχα έλεγε πως ε, εδώ είναι ένα πλούσιο μέρος του κόσμου που έχει ήδη βιομηχανιστεί και τα λοιπά και έχει εκπέμψει τόσους χιλιάδες τόνους και πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω από το 20%. Δεν ξέρω τώρα αν πάμε προς τα πίσω. Με διατυπώσεις που τις έχουμε ψηφίσει τρεις φορές. Ο Καλ Φλόρεντς εδώ πέρα ε, συγκατανεύει. Ελπίζω να μην έχετε παρετηθεί. Έτσι ως κοινοβούλιο πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία και να πούμε πρέπει να είναι πάνω από 20%. Δηλαδή τώρα αν έχουμε 18,4 το 2013 ε, δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να πούμε θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Ακόμα και αν γνωρίζω πως η επίσημη διαπραγματευτική γραμμή είναι πως ε, μετά είναι υπό και με μία σειρά ε, μέτρων όπως το ILOC, ε, τα αέρια ε, τον, τους χλωροφοροανθρακίες και τα λοιπά. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και θα πρέπει νομίζω να κάνουμε κάτι παραπάνω. Το κλιματικό ταμείο είναι άδειο, το είχα πει ήδη, το είπα το πρωί και στον Υπουργό. Χρειαζόμαστε είτε ένα φόρο διοξιδίου του άνθρακα, είτε τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα ήθελα δε να ρωτήσω τον πρόσωπο εδώ πέρα της Κομισιόν αν, υπάρξει κάποια, αν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος όσον αφορά την ομάδα εργασίας για την μέτρηση της, των εκπομπών του διοξιού του άνθρακα για το στόχο των δύο βαθμών, τι σημασία έχουν όλα αυτά για τη Βαρσοβία. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό. Επίσης ε, με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Κόρολετς, έχουμε αυτή τη διαδικασία του ΟΗΕ που πηγαίνει πολύ αργά. Αλλά στον κόσμο συμβαίνουν πολύ περισσότερα. Και μην ξεχνάμε πως υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής των Δημάρχων από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σίδνεϊ συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Τα δηλαδή οι δήμαρχοι τα λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη, κάνουν πράγματα και οι επιχειρήσεις επίσης έχουν δύο πλευρές. Έχουμε τους παλιούς και τους νεότερους που κάνουν πολλά πράγματα από μόνοι τους και νομίζω αυτά τα δύο θα παίξουν μεγάλο ρόλο στη Βαρσοβία. Αυτά ευχαριστούμε για όλα. Ε, κυρία Ντουμπρόβκα. Να με συγχωρείτε. Hvala, <coughs> Είναι ενδιαφέρον να ακούμε τις συζητήσεις γι' αυτό. Πρέπει να δούμε πώς εμείς τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα και να πετύχουμε. Πρέπει να δούμε τώρα πώς θα γεμίσουμε το κενό για να ξεφύγουμε αυτό τον ε, κόσμο τον εικονικό. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω ο προηγούμενος ομιλητής είπε ποιοι θα έπρεπε να συμμετάσχουν. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες χώρες οδηγούν το παιχνίδι, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πότε θα μπορέσει κάτι να προσφέρει στον εαυτό της με 28 κράτη-μέλη. Ναι, εντάξει το σύνολο της Ευρώπης ε, είναι ακόμα μεγαλύτερο πέρα από τις 28 χώρες. Το τέλος του 2009 Ήμουν ε, πρόεδρος ε, σε μια επιτροπή από τις μεγάλες χώρες και την Τουρκία και τη Ρωσία και τον Κάφκασο του Νότου και πολλές περιοχές που δεν συμπεριλαμβανόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε συμμετέχουν σε άλλα όργανα. Αλλά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας αυτά τα κράτη εντάξει μην κάνουμε επαναστατικά ας πούμε αλλά τουλάχιστον η Βαρσοβία και το Παρίσι να μην γίνουν τελικά, να μην καταλήξουν σε καινούρια Κοπενχάγη. Και τώρα για τη συνδιάσκεψη των δημοτικών αρχόντων. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση, αλλά εδώ υπάρχουν και μικρές χώρες, μικρές περιοχές Και νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά. Εμείς μιλάμε πάντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία του περιβάλλοντος. Ε, μήπως αποτελεί μέρος της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και η προστασία της υγείας, ε, το πόσιμο νερό, η εκπαίδευση για επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα αυτά είναι για ανθρώπινα δικαιώματα επίσης. Και οι υπόλοιπε χώρε έχουν δικαίωμα σε ένα υψηλό επίπεδο ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένε ενέργειε και μέχρι το 2015 θα πρέπει να θετήσουμε μια συμφωνία για το κλίμα και να πετύχουμε συγκεκριμένου στόχου για να πραγματοποιήσουμε και αυτά που προβλέπουμε για το 2020. Ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο ξανά στον κύριο Μετσκέρ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, αρκετές ερωτήσεις. Ξεκινήσω με τον κύριο Φλόρεντς, ο οποίος ρώτησε πώς πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμαστεί σε σχέση με το τι μπορεί να συνεισφέρει. Το σχέδιο είναι αρχές του επομένου έτους να έχουμε μια συζήτηση μεταξύ των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι μπορεί να είναι η στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε το οδικό χαρτί 2015, είναι μια αφετηρία, αλλά μας δίθηκε να κάνουμε περισσότερα. Και βεβαίως το θέμα ήταν με το τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να συνεχιστεί αυτή η πολιτική στο μέλλον μετά το 2050 ε, και να αντλήσουμε και τα διδάγματά μας ε, για την εφαρμογή της ε, τωρινής νομοθεσίας. Κάτι το οποίο νομίζω μπορεί να μας φάει άλλο ένα απόγευμα. γνωρίζοντας διαφορετικές απόψεις για την εφαρμογή στην κάθε χώρα. Οπότε απαιτείται χρόνος ακόμα για να δούμε το τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνείς διαπραγματεύσεις. Κάποια κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να λένε κάποια πράγματα, μπορεί να έχετε δει. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναφέρει την θέση του και λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πάει στο 30% των 2050 με, και με μια επιπλέον προσφορά να μειώσει περαιτέρω μέσω πιστώσεων. Υπήρχε ένα άλλο ερώτημα που έλεγε το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, για να ενισχύσουμε τη συμμαχία μας με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αφρικανικές χώρες, μικρές νησιωτικές χώρες. Αυτή τη στιγμή Υπάρχει μια μεγάλη διάσκεψη, είναι πολλοί από αυτούς τους εκπροσώπους αυτών των χωρών στις Βρυξέλλες και συζητάμε το πώς ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας επί τόπου. Νομίζω πως ε, στον κοινοτικό προπολογισμό τα βασικά νούμερα έχουν οριστικοποιηθεί, οπότε πρέπει να δούμε τώρα το τι μπορεί να γίνει στρατηγικά για μια παγκόσμια κλιματική συμμαχία έχοντας κατά νου αυτές χώρες. Θα δείτε πως ε, πολλούς από αυτούς τους που είναι εδώ πέρα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε πρακτικά ζητήματα. Και αυτό είναι άρα και το θέμα της αξιοπιστίας. Δεν διαπραγματευόμαστε μόνο. Αλλά θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα παραδοτέα, κάποια απτή συνεργασία Κάτι το οποίο βεβαίως ε, θα πρέπει και εμείς να μπορούμε να προσφέρουμε κατόπιν για τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Σε δύο εβδομάδες ε, θα δημοσιεύσουμε την επόμενη έκθεση πρόοδου και νομίζω πως ένα νούμερο ήδη αναφέρθηκε το πως έχουν πέσει ακουμπές στην Ευρώπη κάτι το οποίο ξεκάθαρα λέει πως ε, νομίζω πως κάνουμε περισσότερα από όσα είχαν προσχεθεί στην πρώτη περίοδο δεσμεύσεων ακόμα και αν μέρος ε, αυτής της μείωσης οφείλεται στην οικονομική κρίση. Τέλος πάντων είχαμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που είχαμε υποσχεθεί. Δεύτερον, είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί μέχρι το 2020. Οπότε νομίζω πως είμαστε αξιόπιστοι ως προς αυτό. Και σχέση με τις νομοθετικές προτάσεις που συζητιούνται ακόμα, στο Κοινοβούλιο και το Συμβουλίο μπορεί να δώσει λίγο περιθώριο για να καταλήξουμε σε κάποια πιο φιλόδοξα αποτελέσματα του χρόνου. Μετά, μία ερώτηση. Οι συζητήσεις στη Βόνη προσφάτως, όπου μία ομάδα δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις λόγω διαφωνίας για την ημερήσια διάταξη. Αυτό ήταν μετά την Τόχα. Όσοι ήσασταν θα θυμάστε πως είχαμε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τρία λεπτά και 20 δευτερόλεπτα όπου αναφέρθηκαν με μεγάλη ταχύτητα όλες οι μεγάλες αποφάσεις που είχαν ε, και όσο το βλέπατε από το ίντερνετ θα είδατε πως ήταν ένας άνθρωπος στεκόταν μπροστά του και προσπαθούσε να τον ε, εμποδίσει να λάβει αυτές τις αποφάσεις. Και αυτό βεβαίω προσπαθούσε η Ρωσία και εξ ονόματος της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας να τον εμποδίσει να κάνει κάτι τέτοιο. Για να μην υιοθετηθεί δηλαδή κάνει ημερήσια διάταξη. Εν τω μεταξύ είχαμε επαφές ε, η Προεδρία επίσης με την Ρωσική Ομοσπονδία για να λυθεί το ζήτημα πριν συνεδριάσουμε στη Βαρσοβία. Και ελπίζω να συμβεί αυτό έτσι ώστε οι ομάδες αυτές και για την παρακολούθηση, επαλήθευση και την προσαρμογή να συνεχίσουν να δουλεύουν στην Βαρσοβία και να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, αλλά δεν θα έλεγα πως ακόμα είναι 100% σίγουρο κάτι Ξέρετε πως είναι διαπραγματεύσεις. Για τη διαδικασία του ΟΗΕ νομίζω πως είναι σωστό να πούμε πως συμβαίνουν πολλά πράγματα εκτός κυβερνήσεων. Αν δείτε το σύμφωνο των δημάρχων ή τους G40, νομίζω οι 40 μεγαλύτερες πόλεις παγκοσμίω. Και προσπαθούμε να κάνουμε μόνοι τους κάποια πράγματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. πιέζουμε για να πούμε πως πρέπει με κάποιο τρόπο να αναγνωρίσουμε το τι θα κάνουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Αλλά αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί οι άλλοι λένε κοιτάξτε, ε, άρα δεν χρειάζεται καμία δράση από τις κυβερνήσεις. Έχουμε το σύμφωνο των δημάρχων. Γιατί να δεσμευτούμε άλλο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η αναγνώριση είναι το ένα, αλλά δεν μπορεί να αναγνωρίσει, να αντικαταστήσει τη δράση των κυβερνήσεων. Δεν τίθεται ζήτημα υποκατάστασης, παρά μόνο συμπλήρωσης. Ευχαριστώ. Vielen Σας ευχαριστώ. Έχουμε δουλειά μπροστά μας κύριος Υπουργός. Είδε πολύ θετικά το μέλλον. Οπωσδήποτε η αποστολή μας στη Βαρσοβία θα είναι να συνηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερες ΜΚΟ, επιχειρήσεις, ενώσεις, αλλά πριν στείλουμε τη δική μας αντιπροσωπεία Αναμένουμε βέβαια στην υιοθέτηση του προφορικού ερωτήματος προς ε, Συμβούλιο και Κομισιόν. Ποιος θέλει, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι. Όποιος είναι υπέρ του, της προφορικής ερώτησης. Κατά. Κανείς. Ομόφωνα. Σας ευχαριστώ. Στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε ορίσει την προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε στις 10 Οκτωβρίου στην ΕΝΒΗ και θα έχουμε και την ε, ψηφοφορία 21 με 24 Οκτωβρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι πράσινες υπόδομες, ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης. πριν ε, εξαφανιστούν όλοι, θα ξεκινήσουμε με τη προφορική ερώτηση. Λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ωραία. Θα δώσω τον λόγο τώρα στους συντάκτες. Κύριος Ταταρέλα, παρακαλώ. Cari colleghi, Αγαπητοί συνάδελφοι, πλήρως συμμερίζουμε και το περιεχόμενο του κειμένου του ψηφίσματος και της ε, ερώτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Αυτές οι πράσινες υποδομές είχαν και έχουν σημαντικότατο ρόλο για το μέλλον του σχεδιασμού του εδαφικού και για την προστασία του φυσικού ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Στις πόλεις σημαντικότατο ρόλο μπορούν να βοηθήσουν για να βοηθήσουν στη βελτίωση των διαφόρων περιοχών και να προλάβουν ε, ε, πλημμύρες και επίσης ε, για το φυσικό περιβάλλον, δάση, λιπέθρο και να προστατεύσουν τα οικοσυστήματα στην Ευρώπη. Μπορούν να παίξουν έναν τρομερό λόλο για καινοτομία στην πράσινη υποδομή για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και να βοηθήσουμε τις ε, επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουμε ε, τα ειδικά προγράμματα από πλευράς Ευρώπης για τη χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων και επίσης ε, τις πράσινες υποδομές θα πρέπει να συνωματώσουμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης ε, και στην ΚΑΠ ε, για μια υποδομή πράσινη. Σημαντικό είναι μια προσέγγιση σφαιρική για την όλη διαχείριση του χώρου. Θα πρέπει επίσης στην όλη δημιουργική διαδικασία να συμμετάσχουν και όσοι χρησιμοποιούν αυτή την υποδομή, κυρίως οι πολίτες αλλά και τοπικοί φορείς, οι ενώσεις, οι οργανισμοί, οι πολιτικοί, οι ιδιώτες. Θα μπορούν έτσι με την ευθύ να αναλάβουν την ευθύνη τους για την πραγματοποίηση αυτής της υποδομής. Καταλήγοντας, αυτή η πράσινη υποδομή αποτελούν μια άριστη επένδυση που μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομία και στο πρασινό και το μέλλον της Ευρώπης και εκεί μέσα περιλαμβάνεται μια υφόρο ανάπτυξη με λύσεις οι οποίες να έχουν πραγματικά σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσεως. Ευχαριστούμε κύριε Ταταρέλα. Και τώρα, Στέλλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, και εμείς συμφωνούμε με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, και με την διατύπωση της ερώτησης θεωρούμε ότι η αξία των αγαθών που μας προτείνει η φύση υποτιμάται συστημητικά και στην Ευρώπη εξακολουθούμε να επιτρέπουμε να, την υποβάθμιση του φυσικού μας περιβάλλοντος, φυσικής μας κληρονομιάς ε, που μακροπρόθεσμα ε, καθιστά τη φύση ευπαθέστερη με σοβαρές περιβαλλοντικές κρίσεις ε, που όλοι γνωρίζουμε. Ε, οι πράσινες ε, υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα, γιατί πάνω από 60% των πολιτών της Ένωσης ε, διαβιούν σε τέτοια αστικά περιβάλλοντα και επιφέρουν ωφέλη για το άτομο και για την κοινότητα, ωφέλη πολλά και διαφορετικά. λύσεις ε, που βλέπουμε μέσα στην ε, πρόταση όπως τα πράσινα δίκτυα μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Ε, άλλα μέτρα σχετίζονται με το καθαρισμό των λιμάτων, την, τον καθαρό αέρα, την προστασία του εδάφους. Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά τις προτάσεις, δεν χρειάζεται να τις απαριθμώ εδώ. Πιστεύω πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλεται η πρόταση αυτή μέσα από τη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει εδώ, αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει με ποιο τρόπο θα προβάλλει ε, και θα προωθήσει την ανάπτυξη πρασίνων υποδομών στην Ευρώπη, κυρίως σε σχέση με τα μέτρα που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθεί μια πραγματική πολιτική των πρασίνων υποδομών στο πλαίσιο του επομένου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα θέλαμε επίσης να μας διευκρινίσει με ποιο τρόπο αυτή η πολιτική θα μπορούσε να είναι πιο ολοκληρωμένη σε όλους τους τομείς παρέμβασης και σε σχέση με όλα τα διαθέσιμα ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαλεία βάσει και της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή στην πράξη πώς θα υλοποιηθούν αυτά θα είναι σημαντικό να μας το διευκρινίσει η Επιτροπή παραδείγματος χάρη για την προώθηση ε, της ανάπτυξης ε, των πρασίνων ε, υποδομών και η διασύνδεση με το δίκτυο Natura 2000, η βελτίωση της διασύνδεσης των κόμβων του δικτύου, μια σειρά από ερετήματα που περιμένουν απάντηση πώς θα ενταχθούν τα μέτρα στη διαρθρωτική πολιτική, στην πολιτική συνοχή, πώς θα συνδεθούν με τα μέτρα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, τη γεωργική πολιτική, την πολιτική ε, πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και πώς θα διασυνδεθούν όλα αυτά με τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μία, ε, έναν απολογισμό, μία έκθεση υπεπραγματικής να ξέρουμε τι έχει ήδη επιτευχθεί σε αυτό το τομέα και επίσης ως προς το χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξέρουμε τι θα χρειαστεί για να υποστηρίξουμε όσους προωθούν τα σχέδια πράσινης ανάπτυξης ε, για την περίοδο μέχρι το 2014. Ε, υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα που γνωρίζουμε, δηλαδή ε, παραδείγματα πρασίνων υποδομών, όμως καλό θα ήταν να ενισχύσουμε την συνοχή όλων αυτών των επιμέρους προγραμμάτων μέσω μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής ε, που θα είναι τέτοια ώστε να μας επιτρέψει στο έπακρον να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό όλων αυτών των λύσεων, να μην έχουμε κατακαιρματισμένα προγράμματα. Πρέπει να επικρατήσει συνοχή και να ε, διασυνδεθούν όλα αυτά τα επιμέρους προγράμματα και μέτρα. Σας ευχαριστούμε. Γιάν Γκερμπράντι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια έκφραση στα Ολλανδικά. Στο... Στις δύο πίτσες η μία δώρο Το καλό με, την, ε, με τις πράσινες υποδομές είναι ότι πληρώνεις μία και παίρνεις ε, δεν 4 4-5 τώρα. Αν ήταν προϊόν στα μαγαζιά θα έτρεχε ο κόσμος ε, να τα αγοράσει, θα γινόταν χαμός. Αλλά εδώ πέρα είναι δύσκολο να εξηγήσουμε ποια είναι τα ωφέλη. Στις πόλεις αν επενδύει κανείς στο πράσινο έχει Ε, είναι πιο ευχάριστη ζωή, είναι πιο δροσερό το καλοκαίρι. Και οι τιμές των σπιτιών ακόμα ανεβαίνουν. Καλό είναι να όταν κάποιος έχει σπίτι είναι καλό για την κοινωνία, για την κοινωνική συνοχή και το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Να δώσω ένα παράδειγμα στον Άι Μέγγεν. Μπορούσαν να ελέγξουν μεταξύ ενό γκρίζου και πράσινου σενάριου. Υπολόγισαν το κόστος και το όφελος. Με το γκρίζο το λεγόμενο σενάριο έχαναν 225 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με το πράσινο κέρδιζαν 230 εκατομμύρια ευρώ. Μισό, σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ μόνο με το να επενδύσουν σε πράσινες υποδομές. Στην καθημερινή ζωή δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, Όσον αφορά την ενσωμάτωση της, ε, των πράσινων υποδομών στα υπόλοιπα θέματα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη γεωργική πολιτική, τα διαρθρωτικά ταμεία κτλ. Το άλλο σημαντικό θέμα, και αυτό βεβαίως θα είναι ένα ερώτημα μου προς την Κομισιόν, είναι το πώς ε, σκοπεύει η Κομισιόν να μεταφράσει τις ιδέες ε, που έχει ε, σε μια διευκόλυνση για τοπικές, εθνικές και περιφερειακές αρχές να τα χρησιμοποιήσουν αυτά. και αν σκοπεύει να βγάλει νέες κατευθύνες γραμμές για να βοηθήσει ειδικά τις ΟΤΑ για να εφαρμόσουν αυτές οι ιδέες. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε την αρχή του ότι δεν θα υπάρξει κάπου κάποια απώλεια Κοινοβούλιο, Κομισιόν και ίσως και το Συμβούλιο από ό,τι φαίνεται. Καλό είναι λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία και να δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή στο θέμα των διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή έργα υποδομών σε γενικές γραμμές δεν ωφελούν το περιβάλλον, τη φύση, αλλά με κάποιες προσαρμογές μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή αυτή του ότι δεν θα υπάρχει κάποια απώλεια. Οπότε το ερώτημά μου προς την Κομισιόν θα είναι είναι διατεθειμένη να το εφαρμόσει και στις άλλες ε, πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Τέλος η κυρία Άννα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ομάδα σκέφτεται για μια στρατηγική στα πλαίσια των υποδομών που να είναι πραγματικά χρήσιμη. Κατά την ομάδα μου αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή. Να μην είναι όλες οι αρμόδιότητες στην Επιτροπή, αλλά είναι κατενεμένες ε, ισορροπημένα. Χαιρόμαστε που γι' αυτό ακριβώς ε, γίνεται προσπάθεια για μια καλή στρατηγική και επίσης υπάρχει μια κάλυψη των διάφορων πολιτικών. Όσον αφορά την οικονομική πτυχή του όλου σχεδίου, θεωρούμε ότι ειδικά καλό θα ήταν να χρηματοδοτηθεί μέσω ταμείων που υπάρχουν ήδη. Χωρίς ε, να σκεφτεί κανείς να προχωρήσει σε σύσταση νέων, νέες προτάσεις για νέα κονδύλια που είναι δύσκολε και αλλιώς να τα πάρει κανείς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η σκέψη δεν είναι για νέα νομοθεσία ευρωπαϊκή αλλά για να χρησιμοποιηθούν μόνο τα υπάρχοντα ήδη εργαλεία είναι κάπως σπάνιο αυτό. Άρα λοιπόν χαιρόμαστε που η απόφαση που λαμβάνεται είναι να εφαρμοστούν αυτά που ισχύουν ήδη, που υπάρχουν ήδη, παρά να ξεκινήσουμε με νέα. Όπως έλεγα, χρειάζεται καλύτερες πρακτικές ε, και η πείρα των κρατών μελών να χρησιμοποιηθεί ώστε να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα τα διάφορα κονδύλια και να διδαχθούμε από τις εμπειρίες των υπολείπων χωρίς κάθε φορά να προσπαθούμε να επινοήσουμε τον τροχό. Χαίρομαι γιατί φτάσαμε σε μια πολύ σημαντική απόφαση για τις πράσινες υποδομές. Σας ευχαριστούμε. Τώρα να δώσω λόγο στην Κομισιόν κύριο Βαντ που Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους αξιότιμους βουλευτές για τα σχόλια που έκαναν ήδη για την προτιμνόμενη στρατηγική για τις πράσινες υποδομές. Είμαστε ευγνώμονες για το σχέδιο ψηφίσματος που καταθέτεται. Θεωρούμε ότι το follow-up, η συνέχεια που θα δοθεί ε, ως επιτοπλίστων καλύπτεται και από το δικό σας ψήφισμα. Οπότε σας ευχαριστούμε. Για τις πράσινες υποδομές ε, θα ήθελα να τονίσω ότι μόνο και μόνο το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή μια τέτοια πρωτοβουλία είναι ένα ηχηρό μήνυμα για τη δέσμευση που αναλαμβάνουμε Εξάλλου αυτό καταδεικνύει και τη σημασία της ατζέντα σε σχέση με άλλες πολιτικές ε, και θα ήθελα να το τονίσω, δηλαδή αναγνωρίζεται επίσημα ότι υπάρχει πλούσιο δυναμικό στον τομέα των ε, πράσινων υποδομών και πρέπει να το κεφαλαιοποιήσουμε τους επόμενους μήνες και χρόνια για να κάνουμε τη διαφορά ε, ως προς την εκπλήρωση των ευρύτερων στόχων μας για το περιβάλλον και για, την απασχόληση. Δηλαδή είναι πολλαπλά τα ωφέλη αυτής της στρατηγικής και αυτό το τένισαν και όσοι παρενέβησαν στη συζήτηση. Ε, τώρα, ε, αυτά που θα κάνουμε εμείς ε, στη συνέχεια, ξαναλέω, υπάρχουν ήδη διεξοδικά στην ανακοίνωσή μας, θα ήθελα να επιμείνω σε κάποια σημεία που θίξατε κι εσείς. Καθεντεφιμπρίες γραμμές. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα τις εκπονήσουμε και τις επεξεργαζόμαστε τώρα με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως είχαμε εξαγγείλει και στην ανακοίνωση. Σε ορισμένε περιπτώσει έχουμε μάλιστα ήδη δημοσιεύσει κατευθυντήρε γραμμέ για τη διεπαφή, παραδείγματο χάρη με την, ε, τα διευθυντικά, τα περιφερειακά ταμεία. Και τώρα εκπονούμε και άλλε ε, κατευθυντηρίε γραμμέ που ευελπιστούμε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο του τρέχοντο, ώστε τα κράτη-μέλη και όλες οι εμπλεκόμενες ε, αρμόδιες αρχές ε, και όλοι οι αρμόδιοι για τα χρηματοδοτικά μέσα που συνδέονται με αυτή την πολιτική να κάνουν τις σωστές επιλογές για την υποδομή. Είναι ισχυροί μας που έχουμε αναλάβει. Αλλά δεν είναι μονόδρομος, είναι αφίδρομος. ο συλλογισμός μας και ο τρόπος που κινούμαστε. Δηλαδή, τι εννοούμε. Ναι, μεν ναι, έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πράσινες υποδομές ε, με αποδέκτες ε, τα κράτη-μέλη, αλλά αντίστοιχα θέλουμε δέσμευση των αρμοδίων αρχών ε, και διαβεβαίωση ότι και για αυτούς είναι προτεραιότητα οι πράσινες υποδομές. Αν δεν υπάρχει ζήτηση σε επίπεδο κράτους μέλους, λίγα μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χοντρικά. Λοιπόν, με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που κάνουμε αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο κρατών μελών ε, και εξάλλου η ρίστα παρόδο είναι επίκαιρο το να περάσουμε αυτό το μήνυμα στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές ότι αν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία θα χάσουμε την επόμενη εφταετία. Ε, πολύ επιζήμιο αυτό για τις πράσινες υποδομές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας τώρα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, αλλιώς ξαναλέω θα χάσουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ε, ως προς τις ε, δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν, ε, υπάρχουν όπως σας είπα και στα έγγραφα που έχουμε υιοθετήσει. Στα πλαίσια της διαδικασίας της περιφερειακής πολιτικής παραδείγματο χάρη ή στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτική, υπάρχουν ε, ε, ανοίγματα ε, για τι πράσινε υποδομέ, για τη χρηματοδότηση και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ορισμένε φορέ πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στι διάφορε εναλλακτικέ και άρα και πάλι εκεί έχει σημασία η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Και για να γίνουν σωστέ επιλογέ, ξαναλέω, πρέπει να έχουμε το feedback από τα κράτη-μέλη και χρειαζόμαστε κλιμάκωση των προσπαθειών για τι πράσινε υποδομέ πριν το τέλο τη προγραμματική περίοδου που τρέχει τώρα. Άλλο ζήτημα είναι η συνεργασία με άλλους εταίρους, με άλλους οργανισμούς για να καταφέρουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Η αναφορά που κάνουμε ε, στην συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό για τις πράσινες υποδομές είναι κάτι υπαρκτό και ε, είναι μία άλλη πιθανή οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε, κυρίως όταν επιθυμούμε να κινητοποιήσουμε εταίρους που μέχρι του δεν έχουν εμπλάκει σε αυτή τη διαδικασία σε μεγάλο βαθμό, κυρίως μιλώντας ε, για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί και εκεί υπάρχει δυναμικό στο μέτρο που θα προσφέρουμε και εμείς ε, και κίνητρα αλλά και δικλείδες ασφαλείας για να είναι βιώσιμες και να διαρκέσουν οι επενδύσεις που θα κάνει ο ιδιωτικός τομέας επεξεργαζόμενοι και άλλες ε, συναφείς πρωτοβουλίες που απαριθμούνται στην ανακοίνωση. Δεν θα σας τις επαναλάβω εδώ, αλλά μία νομίζω έχει σημασία και αναφέρθηκε και στην παρέμβαση της κυρίας Εστρέλα, την ε, ε, διασύνδεση, τη συνδεσιμότητα και τη διασύνδεση με το δίκτυο Natura 2000. Ε, πρέπει να διερευνήσουμε ε, τις δυνατότητες για το Project NG στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας έτσι μια σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση του κατακαιρματισμού όλων αυτών των προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας έτσι τη γενικότερη αηφορία των δικτύων και των πράσινων υποδομών που θα επιτύχουμε μέχρι το 2020. Δηλαδή τα συστατικά στοιχεία για να φτιάξουμε πράσινες υποδομές, για να γίνει κάτι απτό, σε σχέση με σήμερα ε, συγκεντρώνονται. Μιλήσαμε για την Ολλανδία, δεν είναι η μόνη. Δεν αντικαθιστούμε, δεν αποκλείουμε κάτι με τις πράσινες υποδομές, ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό που αποκαλούμε στα αγγλικά enabling framework, ε, δηλαδή να φτιάξουμε ένα πλαίσιο όπου προτεραιότητα θα είναι η χρηματοδότηση των πρασίνων υποδομών και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε την ένα υποστήριξη του Κοινοβουλίου και ε, συνεργασία με, άλλους, ε, με άλλα θεσμικά όργανα, κυρίως η Επιτροπή των Περιφερειών και ΟΚΙ, γιατί μία διάσκεψη θα διοργανωθεί το Δεκέμβρη για αυτό το ζήτημα, οπότε, α, και να μην ξεχνάμε και το Συμβούλιο, διότι όταν μιλάμε για ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, μπορεί να γίνουν επιλογές που θα είναι υποφελείς ε, για το εγχειρήμα των πράσινων υποδομών. Αυτά ήθελα μόνο να προσθέσω, σχέση με αυτά που ήδη ακούσαμε. Πολύ σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. 24 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. 17 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και από ό,τι φαίνεται ελπίζουμε Νοέμβριο να πάμε στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ όλους όσους συζήτησαν, όσους στήριξαν την ερώτηση, όσους έμειναν μέχρι τέτοια ώρα, τους συναδέλφους, τις συναδέλφους. Καλό σας απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε 25 Σεπτεμβρίου. 9 με 12.30 και 3 με 6.30 και 26 Σεπτεμβρίου 9 με 12.30 και παρακαλώ γράφτε στο ημερολόγιο σας πως στις 26 μεταξύ 3 και 6.30 θα έχουμε κοινή συζήτηση με την Ήτρε αυτά. Καλό σας απόγευμα και σε όσους επιστρέφουν καλό ταξίδι.